ο Τούσκο είναι σε, εκλογική, σε προεκλογική εκστρατεία. Δεν είναι αλήθεια. Ο κύριο Τούσκο προετοιμάζει τη διάσκεψη κορυφή για την ανατολική εταιρική σχέση που θα λάβει η χώρα αύριο στη Ρήγα. Meine... Was rufen die Αγαπητοί συνάδελφοι, ε, να διευκρινίσουμε κάτι. Κύριε Γιούρεκ, το Συμβούλιο εκπροσωπείται από την εκάστοτε Προεδρία. Δηλαδή η παρουσία της ε, κυρίας Υπουργού σήμερα το πρωί είναι κάτι το απόλυτα φυσιολογικό. Για να ε, ξέρετε και καλύτερα, ο κύριος Τούσκα είναι πρόεδρος του, Συμβουλίου και αυτό είναι ε, κάτι τελείως διαφορετικό από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Λοιπόν, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, μας ε, ενημερώνει μετά τη συνάντηση κορυφή και εδώ έρχεται ο κύριος Τούσκ. Βεβαίως ε, θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτό που είπατε δεν είχε καμία απολύτω σχέση με την προεκλογική εκστρατεία στην Πολωνία. Το καταλάβαμε. Πάμε λοιπόν τώρα στην εκλογή αντιπρόεδρου. Σύμφωνα με τα άρθρα 15, 17 και 20 του κανονισμού μας ε, έχω λάβει τις εξής υποψηφιότητες ο συνάδελφος κύριο Φάμπιο Μάσιμο Καστάλντο που δέχτηκε την υποψηφιότητά του και προτέθηκε επίσης και αυτή δέχτηκε η κυρία Άνελη Γέτεν Μέκη. Οι δύο υποψήφοι μου ανακοίνωσαν ότι όπως σας είπα προτάθηκαν και δέχθηκαν την υποψηφιότητα τους. Και η εκλογή θα γίνει με μυστική ηλεκτρονική ψηφοφορία. Για να εξοικειωθείτε λιγάκι ε, με το ηλεκτρονικό σύστημα θα κάνουμε μια δοκιμαστική εκλογή. Όταν θα ξεκινήσει η ψηφοφορία, κυρίε και κύριοι, η οθόνη θα δείχνει το τι ψηφίζουμε. Δηλαδή, ε, θα ψηφίζουμε για τον υποψήφιο, ε, τον κατάλογο των υποψηφίων ε, και εσείς θα πρέπει να πείτε ποιον προτιμάτε πατώντας ε, το μπλε κουμπί και μπορείτε το κουμπί να το πάτε προς τα πάνω προς τα κάτω είναι ο cursor και εάν θέλετε ή βρήκατε τον υποψήφιο που επιθυμείτε εκεί θα πατήσετε το συν Αυτό το ρώτησαν πάρα πολύ. Αν θέλετε να δηλώσετε αποχή, διότι έχουμε δύο υποψηφίους, να πατήσετε το κουμπί που λέει αποχή. Είναι το μεσαίο κουμπί. Και στην περίπτωση αυτή, ναι μεν θα ανάψει το μπλε λαμπάκι, αλλά παρόλα αυτά εσείς θα έχετε συμμετάσχει στην ψηφοφορία δηλώνοντας αποχή. Είναι δυνατό να γίνει αυτό. Και βεβαίως μπορεί να μην θέλετε να συμμετέχετε στην ψηφοφορία. Αυτό είναι δική σας απόφαση. προς ε, μεγάλη σας έκπληξη θα προτείνουμε για άλλη φορά δοκιμαστικά την Μονσέρα Καμπαγέ και η Γιουμίλια Τζόνσον αυτοί οι δύο ε, υποψήφοι έτσι ενδεικτικά για να κάνουμε τη δοκιμή προφανώς. Ξεκινάμε λοιπόν με τη δοκιμαστική ψηφορία. Ψηφίστε, ψηφίστε τι θέλετε από τις δύο που σας ανέφερα. Βλέπετε λοιπόν στην οθόνη σας εμφανίζεται ε, election test. Θα ψηφίστε είτε την κυρία Μονσερά Καμπαγέ είτε την κυρία Μικέλε Τζόνσον. Μπορείτε να κουνήσετε τον κέρσορα προ τα πάνω ή προ τα κάτω και όσοι από όποιον θέλετε, όποιον προτιμάτε, θα κουνήσετε τον κέρσορα και αφού το βρείτε το όνομα και είναι κόκκινο, εκεί θα πατήσετε. Λοιπόν, ψηφίζουμε δοκιμαστικά. Δοκιμαστικά ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Ψηφίσατε όλοι. Ψηφίσατε όλοι παρακαλώ. Έκλεισε λοιπόν η ψηφοφορία. Λοιπόν, η κυρία Καμπαγέ, η Μονσερά Καμπαγέ κέρδισε αυτήν την εκλογή με 309 ψήφους. Check. <laughs> Κύριε Λούκα, θέλετε κι εσείς να δηλώσετε υποψηφιότητα. Παρακαλώ. Όχι, εγώ δεν θέλω να θέσω υποψηφιότητα, αλλά θα ήθελα οι δύο υποψήφοι να ε, συστηθούν λιγάκι, γιατί εγώ τη δεύτερη υποψήφια ούτε που την ξέρω. Κοιτάξτε κύριε Λούκα, δυστυχώς αυτό δεν προβλέπεται στο καταστατικό μας. Οι εκλογές γίνονται χωρίς...